Συμβουλίου θα ε, υπογράψει βάσει του άρθρου 74 του ιστορικού κανονισμού και βάσει της διαδικασίας της, ε, της συνήθους νομοθετικής διαδικασίας ε, νομοθετικές πράξεις που επίσης θα συναυτούν στα πρακτικά της σημερινής συνεδρίασης και τέλος και το εννοώ τέλος βάσει του άρθρου 216 του εσωτερικού κανονισμού οι επιτροπές που είναι αρμόδιες για διάφορα διορθωτικά κείμενα